οι δηλώσει του Συμβουλίου και τη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Εξ ονόματος του Συμβουλίου να δώσω το λόγο στην κυρία Καλνίνα Λούκασέβικτσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ γιατί καλέσατε το Συμβούλιο να συμμετάσχει σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση για το ΕΤΣΕ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Είναι καθεαυτό μια καλή αρχή για περαιτέρω συζητήσεις. Χαίρομαι για την ευκαιρία αυτή να σας εκφράσω τις απόψεις μου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε σημαντικό ρόλο για να έρθει στο προσκήνιο ο ρόλος των επενδύσεων και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ σήμερα μπροστά σας τη στιγμή που αρχίζουμε να μιλάμε για την πρώτη φάση του στρατηγικού σχεδίου επενδύσεων. Για μας είναι μεγάλη προτεραιότητα της Προεδρίας μας και είναι λοιπόν ουσιώδες να ενδυναμωθεί η οικονομική ανάπτυξη και να μειωθεί η ανεργία στην Ένωση. Το, η επενδυτική δέσμη στοχεύει να πετύχει τον διπλό στόχο αυτόν και είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι συνομοθέτες να συνεργαστούν στενά και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Βρίσκω χρήσιμο να σας υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ και το Συμβούλιο έθεσαν ε, χρονοδιάγραμμα πολύ φιλόδοξο και υπολογίζουμε και στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να επιτευχθεί. Η τωρινή κατάσταση των επενδύσεων απαιτεί κάποια αντίδραση και γρήγορη. Θέλουμε τα πρώτα σχέδια να εφαρμοστούν ήδη από φέτος. Το Συμβούλιο ήδη άρχισε να εξετάζει τις προτάσεις σε μια ad κομμάδα εργασίας και πολύ τακτικά. Ήδη έγιναν δύο τέτοιες συνεδριάσεις την περασμένη εβδομάδα και η επόμενη προβλέπεται για αύριο. Θέλουμε ήδη το Μάρτιο να έχει συμφωνηθεί η γενική προσέγγιση για να υπάρξει αρκετός χρόνος να εγκρίνει και το Κοινοβούλιο. Πολύ πριν το, τις καλοκαιρινές διακοπές. Το ΕΚΟΦΗΝ θα παρακολουθεί τα πράγματα αλλά και εσείς θα παίξετε σημαντικό ρόλο διότι η πρώτη εντατική ανταλλαγή απόψεων σε υπουργικό επίπεδο έγινε χθες και είμαι βέβαιη ότι το Κοινοβούλιο θα ενισχύσει τις προτάσεις μας και θα έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία γιατί έτσι θα δοκιμαστεί η αμοιβαία μας δέσμευση να υπάρξει ανάκαμψη στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι. Η σημασία του έτσι είναι προφανής αλλά είναι μόνο ένα τμήμα του επενδυτικού σχεδίου της Κομισιόν. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν πόροι για επενδύσεις, αλλά το δεύτερο θεμέλιο είναι, ο δεύτερος πυλώνας, είναι ο καθορισμός ενός Συμβουλευτικού Σώματος για τις Επενδύσεις στην Ευρώπη το οποίο θα βοηθεί στην έβρεση και ταύτιση των καλύτερων δυνατών επενδυτικών σχεδίων ώστε ο ιδιωτικός τομέας να συμμετέχει πλήρως και τα χρήματα να φτάνουν στην πραγματική οικονομία. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ιδιαίτερα τα μέτρα αυτά που συνοδεύουν τις πρώτες φάσεις λειτουργίας του Ταμείου για να πετύχει αυτό το στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο. Παρ' όλα αυτά, το τρίτος του ίσως πυλώνας είναι ακόμη πιο σημαντικός, οι επενδύσεις για το περιβάλλον, για τις ιδιωτικές ιδίως επενδύσεις. Είναι πολύ ευρύτερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε πολλά, πολλαπλά επίπεδα. Από ενωσιακής απόψεως είναι θέμα συμπλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Ορισμένα μέτρα έχουν ήδη ανακοινωθεί από την Κομισιόν, ας πούμε η Ένωση Κεφαλαίου Αγοράς. Θα θέλαμε και τα τρία όργανα να συμμετάσχουν στην εκπόνηση αυτών των σχεδίων για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει κάτι και σε εθνικό επίπεδο για να αφαιρεθούν οποιαδήποτε φραγμή προς τις επενδύσεις και να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητά τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εξετάζουμε πολλές πιθανές τέτοιες πρωτοβουλίες. Το επενδυτικό σχέδιο συμβαδίζει πλήρως με τις προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας, ιδίως για την ανταγωνιστικότητα. Όπως ξέρετε, το σχέδιο δεν στοχεύει στην επίλυση όλων των προβλημάτων της Ευρωζώνης και της Ένωσης. Μακροοικονομικά, σοκ, αποπληθωρισμός, προβλήματα ενεργειακά κλπ. Αλλά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ιδιαίτερα στοχεύει στην ευελιξία ώστε να υπάρξει ανάπτυξη όντως οι επενδύσεις πάνε μαζί με την φορολογική υπευθυνότητα για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δηλαδή η επένδυση είναι μόνο ένα συστατικό. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε όμως τα άλλα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πειθαρχία. Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να συνεργαστούν αποτελεσματικά και γρήγορα για να διασφαλιστεί ότι το νομοθετικό πακέτο διδέσμη θα έχει πραγματικά αποτελέσματα στην οικονομία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία μου. Ο κύριος Κατά είναι εξ ονόματος της Κομισιόν. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, είναι πάντοτε μεγάλη χαρά να βρισκόμαι στο Κοινοβούλιο και να μιλάω για μείζωνα ζητήματα. Όπω σήμερα. Να ευχαριστήσω για τη Λετωνική Προεδρία για την εξαιρετική τη δουλειά και που έχετε βάλει το επενδυτικό πρόγραμμα τόσο ψηλά στι προτεραιότητέ σα. Μόλι δύο μήνε μετά την ανακοίνωση τη φιλόδοξη στρατηγική για την πρόθεση τη ανάπτυξη και τη απασχόληση στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, υποβάλλει σχέδιο πρόταση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Ταμείου Επενδύσεων. Ε, έχουμε πολύ γοργά αποτελέσματα. Εδώ ε, πηγαίνουμε στην καρδιά τη επιθετική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι επενδύσει. Θέλουμε να λειτουργήσουν τα πιο σημαντικά τμήματα τη ευρωπαϊκή οικονομία και να δημιουργήσουμε θέσει εργασία. Θέλουμε ένα διαφανή διάβλο για την επιλογή προγραμμάτων με ένα κομβικό σημείο που θα επιτρέπει στους θεσμικούς, κρατικούς και ιδιώτες επενδυτές να καταρτήσουν από κοινού βιώσιμα προγράμματα που θα ωφελήσουν όλες τις πλευρές. Ένας από τους στόχους του προγράμματός μας είναι ότι με το κάθε ένα από τα μέτρα μας θα αρθεί η ευεβαιότητα για να υπάρξει όλο ένα και περισσότερη ε, ιδιωτική πρωτοβουλία στις επενδύσεις. Πρέπει με τα κράτη-μέλη να δούμε πώς θα καλυφθεί ο κάθε φορέας, πώς τα κράτη-μέλη και οι συνεισφέροντές τους θα ε, ε, υπολογίσουν τι συνεισφορέ του βάσει του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη και πώ θα υπάρχει και ένα σταθερό αντίκτυπο ε, στην απασχόληση και τι θέσει εργασία. Με τι εταιρείε πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει ένα νομοθέτημα που να εξεργά την διακυβέρνηση, την διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στατικών Επενδύσεων με την κατάλληλη τεχνική επεξεργασία και την αποτίμηση της ε, διάρκειας ζωής των, της των προγραμμάτων. Εργαζόμαστε γοργά και στηριζόμαστε σε εσά για μια σωστή πολιτική στήριξη, ώστε να λειτουργήσει γρήγορα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικικών Επενδύσεων στο πρώτο μισό της φετινής χρονιάς. Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ φιλόδοξο. Το Συμβούλιο ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις στις 19 Ιανουαρίου 2015. Η ομάδα εργασίας για το επενδυτικό πρόγραμμα είχε μόλις δημιουργηθεί και είναι σημαντικό οι εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου να ξεκινήσουν ως το δυνατόν συντομότερα. Υπολογίζουμε στους συνομοθέτες για να ε, συμφωνήσουν το κείμενο, τουλάχιστον ως τον Ιούνιο, και να ε, έχουμε κάτι που να λειτουργεί από τα μέσα του 2015 επειδή προχωρούμε γοργά, σημαντικό είναι να έχουμε το χρόνο να εξηγήσουμε με σαφήνεια τι ακριβώς κάνουμε. Ε, γι' αυτό θέλω να δούμε την διακυβέρνηση, ε, το θέμα των εγγύσεων και ε, βεβαίως το κατά πόσον οι συνεισφορές των κρατών μελών ε, κατά πόσο στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη θα μπορούμε να υπολογίσουμε τι συνεισφορέ των κρατών μελών. Εάν θα χρειάζεται η άμεση συνεισφορά των κρατών μελών ή μέσω συγκεκριμένων τραπεζών του. Θα μπορούν να συμβάλλουν σε διαφορετικά τμήματα των προγραμμάτων τα κράτη-μέλη. Συνεισφορέ σε μορφέ ε, κεφαλαίων ε, είναι κάτι που μπορεί να συναποτιμηθεί με την... δεν θα συναποτιμηθεί με τη δημοσιονομική προσαρμογή. Επίσης πρέπει να αναζητήσουμε τις κατάλληλες πλατφόρμες για τις επενδύσεις που θα είναι επιλέξιμες βάσει της ρήτρας για τις πραγματικές επενδύσεις. Ως προς την διαχείριση, την διακυβέρνηση του Ταμείου διαβλέπουμε μία δομή διπλής ταχύτητας η οποία να σχεδιαστεί για να επιτρέψει στο Ταμείο να αρθεί η βεβαιότητα των επενδυτών με την ανάληψη προγραμμάτων υψηλού κινδύνου από ό,τι συνήθως κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερη σημασία, διότι θα πρέπει αυτό το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Ταμείο να προωθεί προγράμματα ώστε οι επενδύσεις να έχουν ροή προς τις χώρες και τους τομείς της οικονομίας μας που περισσότερο το χρειάζονται. Στην πράξη θα οριστεί ε, ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για την καθοδήγηση επιλογής των προγραμμάτων. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα ορίζουν το προφίλ κινδύνου του Ταμείου και τα κριτήρια για την επιλογή των προγραμμάτων. Αυτό το, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει το, ε, τις ανάγκες των εταίρων και της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και στο μέλλον οποιοδήποτε τρίτο μέρος που μπορεί να συμπληθεί και να συμμετέχει ε, με κεφάλαια ε, ώστε να υπάρχει συμμεταχείριση όλων των εταίρων καθώς οι βασικοί συμβάλλοντες προς το Ευρωπαϊκό Στατικό Ταμείο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όλες τις αποφάσεις ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο θα λαμβάνονται με συνένεση. Η Επενδυτική Επιτροπή που θα συναποτελείται από έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα πρέπει να ε, επιλέγει τα προγράμματα που θα πρέπει επίσης να επιλέγονται με τη σειρά τους βάσει της αξίας τους και να περνάνε και από τον έλεγχο της Εθνικής Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή θα είναι ε, ανεξάρτητη και θα πρέπει να επιλέγει κρίσιμα προγράμματα ε, ώστε να υπάρχει και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα τελικά. Θα πρέπει να οριστούν κριτήρια για την επιλογή των προγραμμάτων που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις ε, εγκριθούν τα σχετικά κείμενα και κανόνες αλλά ήδη τα κριτήρια αυτά είναι σαφή. Τα προγράμματα βάσει αυτής της πρωτοβουλίας πρώτον θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα με τη στήριξη που μπορεί να τους παρέχει το έπειτα να είναι όρημα για να λειτουργήσουν σε παγκόσμιο σκηνικό, τρίτον να ε, υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ένα σύστημα που να συνάδει με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες όπως την στρατηγική για το 2020 για την ε, ολοκληρωμένη και ευφυή ε, και βιώσιμη ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Ε, επίσης θα πρέπει τα κράτη να ε, έχουν προγράμματα υψηλότερου κινδύνου αλλά και με δυνατότητα μεγαλύτερης κερδοφορίας από ό,τι τώρα κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα πρέπει το στρατηγικό ταμείο να χρησιμοποιείται μόνο όπου η χρηματοδότηση δεν είναι διαθέσιμη από άλλε πηγέ ε, με λογικού όρου. Η λογοδοσία του Κοινοβουλίου ε, είναι κάτι σημαντικό γιατί το στρατηγικό ταμείο θα είναι πλήρω υπόλογο, θα λογοδοτεί προ το Ευρωκοινοβούλιο και η παρακολούθηση θα βασιστεί σε δύο αρχέ. Πρώτα απ' όλα υποβολή εκθέσεων. Ε, θα υποβάλλονται ε, δις ετησίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία φορά αναέτος προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στοιχεία για τις ε, δράσεις χρηματοδότησης και επενδύσεων του Στατικού Ταμείου. Οι εκθέσεις θα δημοσιεύονται και επίσης θα υπάρχει και υποβολή έκθεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του κανονισμού. Ως προς τη λογοδοσία το Κοινοβούλιο θα έχει το δικαίωμα να οργανώσει ανα πάσα στιγμή ακρόαση με τον ε, εκτελεστικό διευθυντή του Ταμείου για το, τις του. Επίση, ο εκτελεστικό διευθυντή θα έχει νομικέ υποχρεώσει να απαντά ε, ε γραπτός γραπτό ή προφορικό στι ερωτήσει που θα το απευθύνει το Ευρωκοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο επίση μπορεί να ζητήσει υποβολή έκθεση από τρίτο μέρος. Ε, Κυρίε και κύριοι, οι προτάσει που λάβατε σήμερα θα πρέπει να συμπληρωθούν από μια σειρά από μέτρα για να έρθουν οι φραγμοί ε, κατά των επενδύσεων και να δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία αγορά. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό μέρος του επενδυτικού προγράμματος. Είναι ο τρόπος να αλλάξουμε ε, δομικά την Ευρώπη με μακροπρόθεσμα προς τη σωστή κατεύθυνση και να δράξουμε όλες τις ευκαιρίες επενδύσεων. Ε, αυτό το σύνολο δράσεων ορίζεται στο πρόγραμμα εργασιών του 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα υποβάλουμε και περαιτέρω προτάσεις για την Ενεργειακή Ένωση, την ψηφιακή ενιαία αγορά, την Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών και την ε, ε, ενοποίηση της αγοράς για τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Ε, αργότερα μέσα στη χρονιά θα υποβληθούν σχετικές προτάσεις. Αναπομονούμε για την συνεργασία μαζί σας για τα θέματα αυτά. Και να πω κύριε και κύριοι ότι ενώ υπάρχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες στα κείμενα που τώρα σας στείλαμε, πρέπει να τα συζητήσουμε σαφώς και να τα διευκρινίσουμε, αλλά να μην χάνουμε τη σφαιρική εικόνα. Ε, ποιος είναι ο τελικός μας σκοπός. Η κρίση εμπιστοσύνη δημιουργεί δυσκολίε στις επενδυτικές χώρες μπλοκάρει και αυτό ε, ουσιαστικά πλήττει την πραγματική οικονομία. Τα νέα αυτά μέτρα πρέπει να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και οι επενδύσει να ρέουν προ την περιοχή τη Ευρώπη και του τομεί τη οικονομία μα όπου χρειάζεται δημιουργία θέσεων απασχόληση. Είναι πολύ σημαντικό σε πολιτικό επίπεδο να δράσουμε κατεπηγόντω γιατί το χρειάζεται αυτό και η πραγματικότητα της οικονομίας μας. Ε, θα συνεργαστώ λοιπόν στενά με το σώμα σα για να ε, εγκρίνουμε τι προτάσει αυτέ το δυνατόν συντομότερα και να υπάρξει γρήγορα αυτό το στρατηγικό ταμείο. Ε, πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τώρα, ε, εξ ονόματος των ομάδων, οι συνάδελφοι, πρώτος ο κύριος Βίμπερ, για τέσσερα λεπτά εξ ονόματος του ΕΛΚ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε εκπρόσωποι του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, ευχαριστώ για την παρουσίαση του, από τον κύριο Κατάουνεν. Η ομάδα του ΕΛΚ καλωσορίζει την πρόταση της ε, Επιτροπής για το πακέτο ανάπτυξης και επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω ότι είναι σωστό και το πλαίσιο. Όχι χρέος για επενδύσεις, αλλά ε, να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις για να υπάρξουν ε, θέσεις απασχόλησης. Αυτή είναι η ορθή οδός. Ευχαριστώ για την ταχεία παρουσίαση και τις καλές προτάσεις. θα μιλήσω συνάδελφοι από το ΕΛΚΙ για τις λεπτομέρειες. Θέλω να συνδέσω τη σημερινή πρόταση με δύο εξελίξεις που χαρακτηρίζουν την ε, οικονομική κατάσταση και την πολιτική συζήτηση. Αυτό δηλαδή που είδαμε με τις εκλογές στην Ελλάδα την Κυριακή, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα να αναφέρω ότι η νέα αρχή της Ευρώπης που προτείνει ο νέος Πρωθυπουργός ε, δεν θα έχει επιτυχία. Επιτυχία θα έχουμε μέσω των προτάσεων που είπε ο κύριος Κατάνιον, το πρόγραμμα επενδύσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ILO, σήμερα δημοσίευσε στοιχεία που λένε ότι μέσω αυτών των ε, επενδύσεων θα δημιουργήσουμε 2,2 νέες θέσεις εργασίας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, θα είναι πραγματική όθηση για την Ένωση. Έτσι θεωρούν οι εμπειρογνώμονες που ασχολούνται σε αυτό το τομέα. Αγαπητοί συνάδελφοι, γι' αυτό αναφέρθηκα στην Ελλάδα. Γιατί νομίζω ότι πολλά από αυτά που θέλουμε να κάνουμε για επενδύσεις, για να ενισχύσουμε την οικονομία της Ευρώπης, κινδυνεύουν λόγω του αποτελέσματος των εκλογών και της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Τώρα ο κύριος Τσίπρας αναγγέλει ότι θέλει κατάργηση του χρέους. Πώς είναι δυνατόν οι ιδιώτες επενδυτές να κάνουν επενδύσεις όταν παράλληλα οι πολιτικοί στην Ευρώπη λένε ότι δεν θα πληρώσουμε τα χρέη μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, τι έχει να κάνει με την αλληλεγγύη αυτό όταν Εάν περικοπεί το χρέος της ε, Ελλάδας θα πρέπει να πληρώσουν χώρες όπως η Κύπρος 80 εκατομμύρια. Η Ιταλία θα πρέπει να πληρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια. Η Ισπανία θα πρέπει να πληρώσει 6,6 δις. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ιρλανδία 375 εκατομμύρια. Εάν λοιπόν κάποιοι δεν πληρώσουν, τότε θα πρέπει να πληρώσουν όλοι οι άλλοι για αυτούς. Για την Ελλάδα δηλαδή. Είναι αλληλεγγύη η Ισπανία και η Ιταλία και η Κύπρος να πληρώσουν για τα ελληνικά χρέη, αυτό θα οδηγήσει σε σταθερότητα, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε ασφάλεια και σταθερότητα. Θα οδηγήσει σε αστάθεια. Οι υποσχέσει που έγιναν πριν τι εκλογές ότι θα υπάρξουν 11 δι νέα, ε, νέες δαπάνες, αυτό δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές θα έχουν εμπιστοσύνη στη χώρα αυτή. Και ελπίζουμε και παρακαλούμε οι επιτυχίες που κατάφερε μέχρι σήμερα η Ελλάδα, στο σκελισμένο προπολογισμό, ότι έχει ανάπτυξη σήμερα. Ναι, είναι σε δύσκολη θέση, αλλά έχει σημειώσει ανάπτυξη. Αυτέ οι επιτυχίε δεν θα πρέπει να τεθούν εν κινδύνο. Αυτέ οι αριστερέ ριζοσπαστικέ δυνάμει έχουν συνδυαστεί με δεξιούς ε, λαϊκιστές. Στους σοσιαλδημοκράτε, φίλους να θυμίσω ότι στη νέα κυβέρνηση δεν είναι καμία γυναίκα υπουργό. Μόνο άνδρες. Μόνο άνδρε αυτή η νέα κυβέρνηση. Τι έχει να κάνει αυτό με ισοτιμία των φύλων και ισότητα των φύλων. Γιατί θα αναφέρω όλα αυτά στη συζήτηση για τι επενδύσει, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί αυτέ οι εξελίξει είναι πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από το, για το πόσο οικονομική ανάπτυξη θα έχουμε. Και αν δούμε αυτή τη στιγμή πώ εξελίσσεται η Ευρώπη, στην Ιρλανδία έχουμε 3,6% ανάπτυξη, στην Λετωνία 2,6%, στην Ισπανία πέρυσι είχαμε ένα εκατομμύριο νέε θέσει εργασία. Στην Ισπανία, σε όλες αυτές τις χώρες, όπου υπάρχουν κυβερνήσει του ΕΛΚ, όπου γίνεται σωστή πολιτική με προοπτική προ το μέλλον, έχουμε ανάπτυξη και θετικές προοπτικές. Και εμείς ως ΕΛΚ θα διατηρήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν διάφορες ε, ερωτήσεις μπλε κάρτας. Δέχεστε μία μπλε κάρτα κύριε. Μόνο μία. Η κυρία Φων Στόρχ. Κύριε Βέμπα, καλωσορίζετε τα 300 δισεκατομμύρια πακέτο επενδύσεων. Δεν με εκπλήσει αυτό. Αλλά δύο είπατε ότι δεν θα δημιουργηθούν νέα χρέη. Με εκπλήσει αυτό, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα χρησιμοποιήσουμε δημόσιους πόρους και προσπαθούμε να το αυξήσουμε αυτό σε 60 δισεκατομμύρια για να ενθαρρύνουμε τους ιδιώτες επενδυτές. Αυτό είναι δημόσια χρηματοδότηση. Και δεύτερον, είναι σωστό ότι θα δημιουργηθούν 2,2 ναι, εκατομμύρια θέσει εργασία. Τότε γιατί να μην το διπλασιάσουμε, το τριπλασιάσουμε. Και λύσαμε το πρόβλημα τη ανεργία. Τι επενδύσει δηλαδή. Ο Βέμπερ. Θαυμάσιο ο τρόπο αντιμετώπιση των προβλημάτων. Καλό όμω είναι να συμβάλλουν και οι λαϊκιστέ ε, στι λύσει. Η πρόταση που γίνεται δεν θα αυξήσει το χρέο. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδιώτες επενδυτές. Όποιος έχει ε, σωστή οικονομική σκέψη, αυτός είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσει το θέμα. Γι' αυτό η πρόταση του Κατάινεν είναι σωστή. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Η κυρία Γοντρίγκε από πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα έχουμε την ευκαιρία να βγάλουμε συμπεράσματα για τα πρόσφατα, τις πρόσφατες εκλογές στην Ελλάδα. Το σίγουρο όμως είναι ότι χρειάζεται ένα καινούριο πρόγραμμα για την Ελλάδα με συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με, με βάση την δημοσιονομική υπευθυνότητα αλλά και με πραγματική πρόοδο και πραγματικές προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ελλάδα. Αυτή είναι η μόνη δυνατή απάντηση. Γι' αυτό βέβαια χρειάζονται επενδύσεις και γι' αυτό η σημερινή μας συζήτηση είναι πολύ επίκαιρη και πρέπει να τη φροντίσουμε ιδιαίτερα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρουσιάσω εξ ονόματος της ομάδας μου το γεγονός ότι ανησυχούμε ιδιαίτερα με την μεγάλη καθυστέρηση της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού αυτού Ταμείου. Πράγματι ανησυχούμε γιατί οι χώρες μέλη μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει υποσχέσεις για κεφάλαια. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό θα ήταν ουσιώδες για να μπορέσει το Ταμείο αυτό να αυξήσει τη δανειοδοτική του ικανότητα. Δεν πάει καλά τα πράγματα δηλαδή. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εγγύηση του προϋπολογισμού και η συμβολή του δεν αρκεί. Και επίσης ανησυχούμε γιατί ο κύριος Σόιμπλε πρόσφατα είπε, αρνήθηκε μάλλον την πρόθεση της Γερμανίας να συμβάλλει. Αυτό είναι πολύ κακό σημάδι. Αυτά τα, αυτούς φραγμούς πρέπει να τους ξεπεράσουμε. Η Ευρώπη χρειάζεται μαζικές επενδύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ασφαλίσουμε ότι όλες οι χώρες μέλη και εκείνες που έχουν μεγάλο έλλειμμα θα μπορέσουν να συμβάλλουν. Ελπίζω να το καταφέρετε αυτό μέχρι την επόμενη διάσκεψη της Ευρωζώνης. Ο κύριος Καμάλ από τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ πολύ. Οι συντηρητικοί δέχονται το γεγό, την πρόταση αλλά θα και οι επενδυτές που έχουν χρήματα προς επένδυση εμποδίζονται, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, από υπερβολική γραφειοκρατία και πηγαίνουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Απομένως η πρόταση αυτή δεν θα είναι φανάκια και το θέμα δεν είναι το ίδιο το ταμείο αλλά το λεγόμενο, ο λεγόμενος τρίτος πυλώνας. Ένα παράδειγμα. Εγώ συναντιέμαι με πολλούς παγκόσμιους επενδυτές που μου λένε ότι θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη αλλά φοβούνται ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν θα τους το επιτρέψει. Η πραγματική δοκιμή λοιπόν δεν είναι πόσοι αγωγοί οικοδομούνται, αλλά πόσοι επενδυτές θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν η ενωσιακή νομοθεσία να μην τους εμποδίσει. Από τις αρχές του χρόνου πρέπει να πληρώνουν το ΦΠΑ στη χώρα του πελάτη πλέον και όχι στη χώρα της πώληση. Ξέρουμε τι κάνει η Amazon. Αλλά αυτή η νομοθεσία που είναι ομοιόμορφη για όλους εμποδίζει πολλούς όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία ας πούμε. Δεν μπορούν να ελέγχουν όλους τους, τους πελάτες ή όλες τις χώρες μέλη. Δεν υπάρχει εκεί το ίδιο ε, επίπεδο ΦΠΑ. Και τώρα τους λένε ότι ίσως να παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία αν πουλήσουν τα προϊόντα τους. Τι κάνουν λοιπόν, κλείνουν. Υπάρχουν τρόποι να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ας μιλήσουμε για αυτά τα επενδυτικά προγράμματα λοιπόν, αλλά αν είμαστε σοβαροί πρέπει επίσης να καταργήσουμε, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία από τώρα και μέχρι να γίνει αυτό καμία επένδυση δεν θα μπορέσει να κλείσει το χάσμα. Ε, δεν θυμάστε τι έλεγε ο Bob Dylan How many roads does, a man walk down Ε και εγώ ερωτώ πόσες επενδύσεις πρέπει να γίνουν πριν κλείσουν πόσες, επενδύ, πόσες μικρομεσαίες εταιρείες Φοβάμαι ότι όπως έλεγε και ο Bob Dylan The answer my friend is blowing in the wind Δύο φορές Τέλιτσκα Τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπουργέ Αντιπρόεδρε, η πολιτική μας ομάδα θεωρεί ότι το πρόγραμμα αυτό για το επενδυτικό ταμείο είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Ε, η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχετε ε, υψώσει το επίπεδο των προσδοκιών οι τρεις πυλώνες τους οποίους βασίζεται το πρόγραμμα αυτό είναι οι τρεις πυλώνες τους οποίους είναι θέμα εμπιστοσύνης για τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι ε, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ε, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο πυλώνας για την εσωτερική αγορά είναι καθοριστικός. Θα συμφωνήσω, επαναλαμβάνω μαζί σας. Υπάρχει ένα θέμα πάνω στο οποίο εν μέρη διαφωνούμε. Ε, μας δώσατε κάποιες πληροφορίες σε σχέση με τις διαφορετικές αλλαγές και την αιρεσιμότητα Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να το καταστήσουμε αυτό απλούστερο, ιδιαίτερα σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο ε, παρόν μπορούμε να το λάβουμε υπόψη μας απλά. Αν έχει ένα ουσιαστικό πρόγραμμα επενδύσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιβάλλει τουλάχιστον στα κράτη-μέλη να έχουν και τα δικά τους επενδυτικά τέτοια προγράμματα διαφορετικά από αυτά τα οποία έχουν προταθεί μέχρι τώρα γιατί κάποια είναι ενθαρρυντικά, κάποια δεν είναι διόλου ενθαρρυντικά. Ελπίζω λοιπόν να κάνω τις σωστές επιλογές. Θα ήμουν πολύ πιο βέβαιος, θα ένιωθα ασφαλέστερος αν τα θέματα τα αντιμετωπίσουν οι εσωτερικές, οι δημόσιες διεθνικές διοικήσεις των κρατών μελών, να εφαρμόσουν σωστά την νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πάρα πολύ καλά σε ποιους τομείς τα κράτη-μέλη δεν τα έχουν καταφέρει. Ο κύριος Καβάρη είναι πραγματικός φιλελεύθερος και θα συμφωνήσω μαζί του ότι η μείωση της γραφειοκρατίας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και το ε, κατονομάζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι σαν πρόβλημα υπαριθμών 1. Πάντως, στο Εθνικό Επενδυτικό Σχέδιο ή οποιοδήποτε τέτοιο είδους πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα προτινόμενα βήματα. Δύο τελικές παρατηρήσεις και τελειώνω. Θα περίμενα κάπως περισσότερα από τη Λετωνική Προεδρία από αυτά τα οποία παρουσίασε σήμερα. Να μην μας λέγατε μόνο ότι έγιναν κάποιες συναντήσεις όπως αυτές της Δευτέρας. Μας ενδιαφέρει το τι έγινε στις συναντήσεις αυτές, ε, ποια είναι η βασική σας όθηση τι θέλετε να αφήσετε. Αυτό έχει σημασία και πρέπει να μας το δείξετε. Εύχομαι λοιπόν καλή τύχη, θα σας στηρίξουμε, αλλά θέλουμε αποτελέσματα και για τους δύο πυλώνες από πλευρά των κρατών μελών. Το λόγο έχει τώρα ο κ. Παπαδημούλης. Ε, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Βέμπερ, καταλαβαίνω την πικρία σας, γιατί έχασε ο φίλος σας, ο κύριος Σαμαράς, τις εκλογές στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι δημοκρατία. Και σας συμβουλεύω να αφήσετε την κινδυνολογία και τη διαστρέβλωση των θέσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Οι Έλληνες πολίτες ψήφισαν εναντίον μιας καταστροφικής λιτότητας που έφερε τεράστια ύφεση, τεράστια ανεργία, τεράστια φτώχεια και άδικη κατανομή των βαρών γιατί οι πλούσιοι φίλοι σας στην Ελλάδα με ευθύνη των πολιτικών σας φίλων δεν πληρώνουν φόρους. Και αυτό είναι ελπίδα για όλη την Ευρώπη κυρία Πρόεδρε. Το τέλος μιας μονόπλευρης λιτότητας. Και εμείς λέμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ότι είναι ώρα όπως ο κύριος Ντράγκη είπε θα κάνω whatever it takes για να προστατεύσω το ευρώ και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να κάνουν whatever it takes για να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στη θέση της καταστροφικής λιτότητας, ενισχύοντας και με δημόσιους πόρους το ανεπαρκές πακέτο Juncker και με συμβολή των κρατών μελών και του Συμβουλίου και με κριτήρια κατανομής των επενδύσεων όπου οι επενδύσεις να πάνε στις χώρες που υποφέρουν από μεγαλύτερη επένδυση, από μεγαλύτερη ανεργία, από μεγαλύτερη φτώχεια αυτό που έγινε στην Ελλάδα την Κυριακή και ευτυχώς το σέβεται και η Κομισιόν και το Συμβούλιο σε αντίθεση με τον κύριο Βέμπερ ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λούκε επιθυμεί να σας θέσει ερώτηση. Δέχεστε. Κύριε Λούκε. Χωρίς μικρόφωνο. Ο συνάδελφός μου Βέμπερ εξήγησε ότι η Ελλάδα έλαβε αλληλεγγύη από την Ευρωζώνη. Θα συμφωνήσετε ότι από αυτή την αλληλεγγύη δεν έφτασε τίποτα μέχρι τον ευρωπαϊκό λαό, ότι ο ευρωπαϊκός λαός υπέστη τα δεινά της ε, πολιτικής λιτότητας, ότι η ανεργία έχει φτάσει σε απίστευτα ύψη, ότι ιδίως η απεργία των νέων έχει φτάσει στα ύψη, ότι η αλληλεγγύη της Ευρωζώνης κυρίως ωφέλησε τους πιστωτές και τις τράπεζες prise de parole. Η Νέα Δημο... Για όσα περιγράφεται, τιμωρήθηκαν οι φίλοι του κυρίου Βέμπερ, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αλλά η λύση, κύριε Λούκε, δεν είναι η επιστροφή της Ελλάδας στη δραχμή, όπως εσείς προτείνετε, γιατί τότε θα χάσουν τα χρήματά τους και οι Γερμανοί φορολογούμενοι. Η λύση είναι μια στροφή και της Ελλάδας και όλης της Ευρωζώνης στην ανάπτυξη με δικαιοσύνη και με μεγάλες μεταρρυθμίσεις εναντίον του πελατειακού κράτους, εναντίον της φοροδιαφυγής, εναντίον της διαφθοράς που 40 χρόνια Νέα Δημοκρατία και Πασόκ έφτιαξαν στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Euh, Συνεχίζουμε λοιπόν με τις πολιτικές ομάδες για την ομάδα των Πρασίνων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να μιλήσω και πάλι για το επενδυτικό ε, πρόγραμμα και ίσως να αφήσουμε τη συζήτηση για την Ελλάδα για αργότερα. Να ευχαριστήσω καταρχά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επενδυτικό αυτό σχέδιο το οποίο επιτέλους δίνει περιθώριο σε επενδύσεις μετά από τόσες χρόνια α, ε, λιτότητας. Σήμερα λοιπόν έχουμε όμως με το επενδυτικό αυτό σχέδιο τρεις ενστάσεις και με την αντίδραση του Επιτρόπου Κατάινεν. Καταρχάς, ότι δεν υπάρχει επαρκή δημοκρατικός έλεγχος. Αναφέρεται μεν στο σχέδιο ότι στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να συμβάλλει στις γενικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό είναι ασαφές. Αν δούμε από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά, από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Υπάρχει ένα Εποπτικό Συμβούλιο, αλλά πώς θα διαμορφωθεί το σχέδιο. Αυτό που είναι κρίσιμο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει απόλυτα ως νομοθέτης για να αποφασίσουμε πώς θα ε, διοχετεύονται οι πόροι αυτοί κατά δεύτερον. Δεν μιλάμε επαρκώς για το κοινό συμφέρον. Το σχέδιο μιλάει για όλα τα πράγματα. μιλάμε για εκατομμύρια σε, εργοστάσια, άνθρακα, χάλιβα. Ξέρουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε και στο Βέλγιο και στη Φλάνδρα ιδιαίτερως βλέπω και τους συναδέλφους από τη Φλάνδρα. Πώς θα φροντίσουμε αυτές οι επενδύσεις να είναι υπέρ του κοινού συμφέροντος. Τρίτον και συντόμως χρειάζεται να δοθεί όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά τι θα γίνει με την φοροποφυγή και πώς θα αντιμετωπιστεί η χασούρα εισοδημάτων. Σας ευχαριστώ, κύριος Γούλφο τώρα από το EFTT για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κατάιναν, αναγνωρίζω ότι είστε ένας από τους επιτρόπους, ο οποίος αν πολλής κατανοεί την εξαιρετικά κακή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωζώνη. Μετά από την σύγκρουση του 2008 η Ευρωζώνη είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο η οποία δεν έχει ανακάμψει. Οι επιπτώσεις στους λαούς της είναι πολύ σημαντικές. Ανεργία, αυτοκτονίες, λιτότητα και βλέπουμε τι γίνεται και στην Ελλάδα. Οι καλοπροαίρετοι κύριε Κατάινεν θέλουν να βρουν λύσεις. Οι λύσεις όμως τις οποίες αναζητείτε με αυτό το στρατηγικό πρόγραμμα δεν είναι σωστές σε μια απελπισμένη προσπάθεια να κάνετε ό,τι κάνουν και στις Ηνωμένε Πολιτείε, κάποιοι πανεπιστημιακοί βρίσκουν κάποιες εντελώς στρεβλές λύσεις. Εμένουν σε αυτές τις λύσεις, τις προπαγανδίζουν, κάνουν σεμινάρια για το ευρώ, ενώ πρέπει να αναγνωρίζετε ότι τελικά το ευρώ είναι το πρόβλημα. Και άμα μένετε στο ευρώ δεν πρόκειται εσείς με 20 δις να δημιουργήσετε 315. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαριανόπουλος, ένα λεπτό. Πολλοί αχαιρετίζουν το επενδυτικό πακέτο Γιούγκερ και την προσωπική χαλάρωση Δράκη, μα γιατί υπηρετεί αποκλειστικά τα δικά του συμφέροντα στα πλαίσια τη επεκτατική διαχείριση τη καπιταλιστική οικονομία. Είναι δύο μορφέ κρατικών επιδοτήσεων με δισεκατομμύρια για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων που θα πληρώσουν πάλι οι λαοί σαν χρέος με νέα αντιλαϊκά μέτρα. Οι ποικιλώνυμοι υπερασπιστές της Ένωσης που συνοστίζονται για τη στήριξη αυτού του μείγματος αποκρύπτουν τη βασική προϋπόθεσή τους. Παραπέρα μείωση αυτού που ονομάζουν εργατικό κόστος, μεταρρυθμίσεις μισθολογικών και ασφαλιστικών συστημάτων για την ενίσχυση των ιδιωτικών επιδίωσεων, δηλαδή κούρεμα των λαϊκών εισοδημάτων, μεταφορά φορολογίας από την εργοδοσία στους εργαζόμενους, γενίκευση της ευέλικτης εργασίας αυτά θα ψηφιστούν στο επόμενο διάστημα σαν ευρωπαϊκό εξάμεινο. είναι ανάπτυξη για τα μονοπόλια και όχι για το λαό που δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα αλλά να οργανωθεί να αντεπιτεθεί με κριτήριο τα δικά του συμφέροντα τι δικέ του ανάγκε. Σας ευχαριστώ η κυρία Γκοστέτα. Έχει το λόγο ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, Υπουργέ δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε πράγματι ανάγκη από ένα σημαντικό κίνητρο για να βγούμε από αυτήν την ευρωπαϊκή κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατανοήσει για το κατεπήγον της υπόθεσης αυτής. Έχει σημασία λοιπόν στις προτάσεις οι οποίες γίνονται από την Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει το δικό του ρόλο στη διαχείριση του ταμείου αυτού. Συμφωνούμε φυσικά με τις προτεραιότητες οι οποίες έχουν διατυπωθεί. Συμφωνούμε επίσης και για τη δημιουργία μιας διαδικασίας επιλογής των προγραμμάτων διαφανέστερης που θα προσελκύσει τους επενδυτές. Πρέπει όμως να είμαστε ελκυστικοί. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τη γραφειοκρατία να τους κάνουμε να επιθυμήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σωστό μήνυμα ε, είναι σαν παράδειγμα να είμαστε πολύ πιο ε, δημιουργικοί στον τομέα της τεχνολογίας γιατί κάτι τέτοιο θα θέσει σε κίνδυνο τις ε, πιθανότητες ανάπτυξης που έχουμε. Δεν θέλω να θίξουμε το πρόγραμμα Horizon 2020. Το έχουμε πραγματικά πολύ ανάγκη. Έχουμε δώσει σκληρούς αγώνες εδώ στο Κοινοβούλιο εδώ και λίγους μήνες. Τελειώνω Πρόεδρε. Λέγοντας ότι η ευθύνη των κρατών μελών είναι τεράστια γιατί αυτές είναι που καθυστερούν για τη συμμετοχή στο ε, πρόγραμμα αυτό ανάλογα με τα δημοσιονομικά τους. Κύριε Γουλφ, σας δώσαμε το λόγο και θα δώσω το λόγο στην κυρία Τομά για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπουργέ Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Δεν συμμερίζομαι την άποψη αυτών οι οποίοι λέγουν ότι ο κύριος Γιούνκερ είναι ένας ταχυδακτυλουργός και δεν θα τα βρει αυτά τα 300 δις. Νομίζω όμως ότι πρέπει να ονοματίσουμε τα πράγματα με τον σωστό τρόπο. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν δημόσιες επενδύσεις. Αυτό θα πρέπει να φαίνεται και στον κοινοτικό προϋπολογισμό και έτσι τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσουν να ενθαρρύνουν τους ιδιώτες επενδυτές. Η Επιτροπή έκανε ένα πρώτο βήμα το ζητάμε εμεί αυτό από την αρχή της κρίσης. Αυτά τα 300 δις σε τρία χρόνια δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη, αλλά θα τα χρειαζόμασταν σε αιτήσια βάση αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να κινητοποιηθούμε με διαφορετικό τρόπο, κυρίως συνεισφέροντας α, στο ταμείο αυτό. Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια νέα ερμηνεία της έννοιας της ευελιξίας στο Συμβούλιο. Υποσχόμενοι ότι αυτό θα βοηθήσει στην ανάκαμψη των επενδύσεων. Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες όμως σε σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση. Η βιωσιμότητα των προγραμμάτων παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν θέμα που έχει άμεση σχέση με την επιλογή των προγραμμάτων. Όμως το άρθρο 5 αναφέρεται σε θέματα εκπαίδευσης, σε θέματα κατάρτισης, τα οποία είναι επιλέξιμα. Πώς θα υπολογιστεί και θα αξιολογηθεί η συγκεκριμένη αυτή βιωσιμότητα, ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα. Πώς ο στόχος της απασχόλησης θα ληφθεί υπόψη γιατί αν το Συμβούλιο και η Επιτροπή ορκίζονται στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Επιτροπής, πώς θα πάρουν τις αποφάσεις τους οι εμπειρογνώμονες στη συγκεκριμένη Επιτροπή του Επενδυτικού Αυτού Στρατηγικού Ταμείου, σε το μίσο όπως η απασχόληση των νέων, η μετάβαση σε νέες τεχνολογίες κτλ. κτλ. Θα ξαναπάρετε το λόγο. Έχετε μία μπλε κάρτα. Τώρα. Κυρία συνάδελφε, κυρία Τόμα, είπατε ότι ζητείτε κάθε χρόνο δισεκατομμύρια σε επενδυτικά προγράμματα. Δεν λέτε όμως από πού θα χρηματοδοτηθούν αυτά. Δεν λέτε ακόμη ότι η ποσοτική χαλάρωση στο Ενωμένο Βασίλειο ή στις Ενωμένες Πολιτείες συνδυάζεται αυστηρά με διαρθρωτικές προσαρμογές συζητείτε τελικά προγράμματα επενδύσεων τα οποία δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν. Η κυρία Τωμά. Μα νομίζω ότι εδώ συμφωνώ απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που κάνουμε είναι δημόσιες επενδύσεις. Χρησιμοποιούμε τον κοινοτικό προϋπολογισμό ως εγγύηση για μόχλευση άλλων κεφαλαίων. Και με τη νέα ερμηνεία από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Συμφώνου Σταθερότητα, ζητούμε από τι χώρε μέλη να επενδύσουν. Αυτό λέω. Και μια και μου δώσατε λίγο χρόνο παραπάνω, να πω ότι ακριβώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη όλες οι χώρες μέλη να ωφεληθούν από αυτό το Ταμείο Επενδύσεων. Και θέτω το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει διακόπτη η πρόεδρος χτυπώντας το σφυράκι της. Πώ θα καταλήξει τα χρήματα αυτά στις περιφέρειες εκείνες που αντιμετωπίζουν τι μεγαλύτερε δυσκολίε. Κύριε Σταρμπάτη, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διέπεται μια κεντρική φιλοσοφία. Αντιδρά σε κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις με οράματα και με ταμεία. Θυμίζω την στρατηγική της Λισαβόνας. Το 2000 είχε θέσει νέους στρατηγικούς στόχους τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει ο ανταγωνιστικότερος και ισχυρότερος οικονομικός χώρος στον κόσμο και το ευρώ υποτίθεται ότι θα διευκόλυνε την, ε, ε, την επίτευξη του στόχου αυτού. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σωρό από ε, κατεστραμμένα όνειρα. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Καταστρώνει ένα νέο σχέδιο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Όποιος καθίσει να αναλύσει το σχέδιο αυτό αντιμετωπίζει υποθέσεις όπου γνωρίζει ο καθένας που έχει ασχοληθεί με τα πράγματα αυτά ότι εάν αλλάξει έστω και μια από τις υποθέσεις αυτές εργασίας καταραίει ολόκληρο το οικοδόμημα. Ακούστε τι είπε ο Μπρέχτ. Ναι, καθίστε να κάνετε σχέδια. Και ανάψτε ένα μεγάλο φως. Κάντε και άλλο σχέδιο και τα δύο δεν θα αποδώσουν, δεν θα ανάψουν. Ένα μισή λεπτό. Ο κύριος Γνωρίζετε ότι το δεύτερο σχέδιο για την συνοχή διαπιστώνει την υποχώρηση των στόχων συνοχής από το 2008. Ευχαριστώ την προσοχή στο εξή. Εάν τα δισεκατομμύρια των επενδύσεων κατευθυνθούν ιδίως στις πλουσιότερες περιφέρειες, τότε όλα τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής κινδυνεύουν να εξοδετερωθούν και οι ανισότητες μεταξύ περιφερειών να επιδεινωθούν. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν ώστε κάθε κατηγορία περιφέρειας, κάθε είδος περιφέρειας να επωφεληθεί από το σχέδιο αυτό. Δεν είναι απλή ευχή αυτή που διατυπώνω, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση που επιβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επακρυπνεί επίσης ώστε το σχέδιο αυτό να χρηματοδοτήσει όχι μόνο εκείνα τα οποία χρηματοδοτούν ήδη οι βιομηχανίες και έχει, είπατε ότι τη χρειάζεται να αναλάβουμε κίνδυνο και χρειαζόμαστε ένα new deal για την Ευρώπη έρχονται στο μυαλό μου για παράδειγμα επενδύσεις στην οικονομία της θάλασσας επενδύσεις στον πολιτιστικό κλάδο επίσης σκέφτομαι τις περιοχές εκείνες που βρίσκονται σε δυσκολία, όπου έχουν όμως νεαρούς και νεαρές με γεμάτους ταλέντα, ιδίως για τις ε, ψηφιακές τεχνολογίες και τελειώνω με ένα σχόλιο ακόμα για την διακυβέρνηση που είναι βέβαια σίγουρο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίζει ρόλο διότι οι επιλογές αυτές δεν θα είναι άλλο παρά πολιτικές. Ένα λεπτό η κυρία Βάνα. Κυρία Πρόεδρε, η μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας μιλεί για 2,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2018 με το νέο σχέδιο επενδύσεων αλλά υπό την προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα θα γίνουν μαζικές επενδύσεις στην αγορά εργασίας και ιδίως στις περιφέρειες εκείνες όπου σήμερα σημειώνεται πολύ υψηλή ανεργία καθώς και με συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της παιδείας, της εκπαίδευσης και ούτω καθεξής. Βέβαια, ο αντιπρόεδρο Κατάινεν στην Επιτροπή προπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου είπε καθαρά ότι στόχο του σχεδίου επενδύσεων είναι η προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών και η αύξηση της αγωνιστικότητα. Σήμερα, ωστόσο, ακούσαμε τι βασικέ αρχέ τη Ευρώπη 2020 με στόχου περιβάλλοντος, στόχου καταπολέμησης τη στόχιας, κοινωνικού κλπ. Παραμένει γεγονό, ωστόσο, τα κριτήρια αυτά έω τώρα για το σχέδιο επενδύσεων δεν έχουν διατυπωθεί ούτε είναι δεσμευτικά. Ρωτώ, Πώ θα εξασφαλίσετε αυτά τα ποιοτικά κριτήρια να ληφθούν υπόψη ω κατευθυντήρες γραμμέ από το ίδιο το steering board. Ζάνι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το πρόγραμμα επενδύσεων έχει σαν στόχο να γίνει μια ακόμη τραγική αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανίκανης για μια ακόμη φορά να ξεπεράσει την οικονομική κρίση βασίζεται ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά τα ιδιωτικές επενδύσεις. Ενώ η κατάσταση αυτή που επικρατεί σήμερα δεν θα πείσει τους επενδυτές να βάλουν τα λεφτά τους. Μόνο μια μαζική δημόσια διαδικασία επένδυσης μπορεί να επηρεάσει θετικά τα πράγματα. Τα υπόλοιπα όλα είναι μυστικιστικές και ουτοπίες, και διαδικασίες και ουτοπίες χωρίς οι Ηνωμένε Πολιτείε βγήκαν από την κρίση αυξάνοντας το, το χρέος τους αλλά έχουν την τύχη να μην έχουν κανόνες σαν του Μάστριχ που σφάζουν την, την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης να δούμε πώς θα βρούμε και τα 20 δις τα οποία χρωστάμε και να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. Κονσάλες Πόνς, ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Κατάινερ. Εμείς υποστηρίζουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Θα πρέπει να λειτουργήσει με την αρχή της προσθετικότητας, δηλαδή σε καμία περίπτωση να μην αντικαταστήσει τις παρεμβάσεις και τις επενδυτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, να αναλάβει επίσης επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου. Σημεριζόμεθα τους στόχους αυτού του Ταμείου, που θα πρέπει να επηρεάσουν άμεσα την οικονομία και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει να επιλεγούν επενδύσεις υψηλής ποιότητας, υψηλής τεχνολογίας και επενδύσεις που δημιουργούν ε, θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια πάρα πολύ σωστή επιλογή γιατί δεν πρέπει να διαψεύσουμε τις προσδοκίες και θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες οι κυβερνήσεις να προχωρήσουν. Οι κυβερνήσεις πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Μια αλλαγή κυβέρνησης δεν σημαίνει αλλαγή κράτους. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τις οποίες έχουν κληρονομήσει. Συνεπώς λοιπόν αλλιώς θα γίνουμε μια περιοχή υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να μην αυξήσουμε τα επίπεδα κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν τις υποχρεώσεις μας γιατί αλλιώς θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και όχι μόνο η Ελλάδα. Ευχαριστώ κύριε Γκονσάλες Πόνς, έχετε μία μπλε κάρτα διευκρινίζω ότι θα σταματήσουμε τη διαδικασία της μπλε κάρτας γιατί έχουμε ένα πολύ μακρύ κατάλογο Τσάνι ε, θα θέσει το ερώτημα. Κύριε Ζάνη έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο το εξής. Σωστά κατάλαβα ότι αμφιβάλλει σε ό,τι αφορά το ταμείο αυτό. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τα εθνικά ταμεία. Είπα ότι το ταμείο αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψη μια βασική αρχή, την αρχή της προσθετικότητας. Συνεπώς τα χρήματα τα οποία θα προοριστούν προς το Ταμείο αυτό των επενδύσεων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τα χρήματα και τις επενδύσεις και τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είναι πολύτιμα για τις χώρες και τις περιφέρειες. Βαν Μπρέντ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε και Συμβούλιο. Πολλά ακούσαμε για την Ελλάδα και νομίζω ότι η συζήτηση δεν θα πρέπει να γίνει εδώ για την Ελλάδα, αλλά θα μπορούσαμε να, μάθει, να μάθουμε κάτι γιατί από τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τη δημοκρατία, αφενός, κατά δεύτερον ότι όλο και μεγαλύτερη υποστήριξη ε, υπάρχει από τον λαό για μια διαφορετική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Μπορούμε να συζητήσουμε το τι σημαίνει αυτό αλλά χρειάζεται ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Με μεγαλύτερη φιλοδοξία θέλουμε εμεί. Αλλά το γεγονό ότι υπάρχει το επενδυτικό πακέτο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονό ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είναι κρίσιμο. Στι συζητήσει για το μέλλον συχνά αναφέρουμε τι ε, διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Πολύ συχνά το ακούμε αυτό. Εμεί από του σοσιαλιστέ και δημοκρατέ είμαστε υπέρ των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αλλά ποιε διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει χρειάζονται ποιες βρίσκουν τη συνένεση και ποιες είναι οι πιο σημαντικές για το μέλλον. Μία από τις μεγαλύτερες τέτοιες είναι η μεταμόρφωση της οικονομία μας σε μια βιώσιμη πράσινη οικονομία. Γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε και το Παρίσι, το κλίμα. Εκεί θα πρέπει να βρούμε τις μεγαλύτερες ε, συμφωνίες και συνενέσεις και αυτό να ενταχθεί και στο επενδυτικό σχέδιο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο συνάδελφος ε, Μπάς ε, το ανέφερε αυτό και μίλησε για το τεράστιο πακέτο προτάσεων που έχουμε ενώπιόν μας και έχουν γίνει σχετικές ε, αναλύσεις και φαίνεται ότι πάνω από 600, το μεγαλύτερο τμήμα των ετοιμάτων έχουν να κάνουν με την καλή χρήση πηγών ενέργειας. Έχουμε 600 δισεκατομμύρια που έχουν μαζευτεί σε αιτήματα για βιώσιμη οικονομία. Το διπλάσιο από αυτά τα χρήματα που έχουμε. Αυτό θα πρέπει να φροντίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι μόνο να επενδύσουμε, αλλά να επενδύσουμε στο μέλλον με βιώσιμο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ουρτάσον για ένα λεπτό. Εμείς εξεπλάγει από αυτά τα οποία μας είπατε στην Επιτροπή Οικονομικών Προϊόντων ότι δεν υπάρχει καμία δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή ανάληψη υποχρέωσης για τη συμμετοχή στο Ταμείο Juncker ε, και πολύ φοβάμαι ότι αυτό το Ταμείο δεν πρόκειται να ε, κάνει τίποτα, να οδηγήσει πουθενά και θα επηρεάσει αρνητικά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όπως το Horizon 2020 και το Connecting Europe θα πρέπει να υπάρξει μια μελέτη για τις μη επιπτώσεις στα προγράμματα αυτά. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει και αιρεσιμότητα σε σχέση με τα προγράμματα αυτά και για το περιβάλλον και για, την, για το κοινωνικό περιβάλλον. Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αγνοηθούν αυτές ε, οι προσπάθειες που δεν θα πρέπει έτσι και να θίξουν τις αντίστοιχες άλλες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ένα λεπτό κύριε Φερνάντες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί μια καινοτομική προσέγγιση η οποία μπορεί να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης ε, για τις επιχειρήσεις, να στηρίξει την επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο ε, επιχειρηματικό τέτοιο και επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα έχει θετικές ε, επιπτώσεις και θα επηρεάσει θετικά την αγορά εργασίας. Μπορεί να καταργήσει εμπόδια στην ιστορική αγορά. Μπορεί να προωθήσει και να βελτιώσει την ε, δικτύωση των ενεργειακών δικτύων και των ψηφιακών δικτύων. Θα αυξηθεί και η ανεξαρτησία μας από ενεργειακές πηγές και η ανταγωνιστικότητά μας. Χρειάζεται όμως νομιμότητα και διαφάνεια. Θα πρέπει να είναι συμμετοχικά τα έργα αυτά. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλους τους φορείς του εκάστοτε κράτου μέλους και θα πρέπει εντατικά να συμμετέχει στο σχέδιο αυτό το Κοινοβούλιο έχει και έναν συντελεστή αλληλεγγύης, ε, εσωτερικής αλληλεγγύης, ε, περιφερειακής ένταξης στο πρόγραμμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπούλμαν για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Καμάλ δεν έχει πλέον την ευχαρίστηση να συμμετέχει στην ζωηρή μας συζήτηση, αλλά αν ήταν εδώ θα του έλεγα, αφού θυμάται τον Μπομπ Τίλαν, να πει και το, σωστή, και το σωστό στίχο εγώ λέω the times they are changing. Αυτό είναι το μότο των σημερινών ημερών. Χρειάζεται λοιπόν πρώτα πρώτα κάποια κοινή στάση, κάποια ενωμένη στάση. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει πλέον καμία δύναμη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε στην πολιτική Ευρώπη, που να μην δέχεται ότι έχουμε ένα τεράστιο κενό επενδύσεων και ότι καλούμεθα να κάνουμε κάτι και γρήγορα για να επανέλθει η ανάπτυξη, να επανέλθει η απασχόληση. Κυρίε και κύριοι, αυτό νομίζω μας ενώνει όλους. Τεχνικά τίθεται το ερώτημα τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό. Αγαπητέ Αντιπρόεδρε Κατάινεν, εδώ μπαίνουν κάποια ερωτήματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν. Και βεβαίως εμείς συναποφασίζουμε, δόξα τω Θεώ είμαστε εδώ. Πρώτο λοιπόν, κοινοπραξίες δημόσιο ιδιωτικού τομέα. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο από τα χέρια των ιδιωτών και αν πετύχει μοιραζόμαστε τα ωφέλη. Αλλά πώς θα καταφέρουμε να βάλουμε τα χρήματα στα σωστά τετραγωνάκια, εκεί όπου δηλαδή θα δημιουργηθεί μελλοντικά η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Και γι' αυτό απορρέουν από αυτήν την ερώτηση άλλες δυο. Ποιος αποφασίζει για την διακυβέρνηση του νέου αυτού εργαλείου. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει λεφτά, αν έχουμε εμεί τη λεγόμενη ownership, δεν θα αφήνουμε στην καρταρόμπα την ευθύνη για να έλθουμε μετά να συζητήσουμε εδώ. Λοιπόν, για τον τύπο οφείλουμε να συζητήσουμε. Δεύτερο, πρέπει να αναπτυχθεί ποικιλία έργων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μείγμα πολιτικής για τα εργαλεία. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε στη συναπόφαση και θα βρούμε τρόπους, είμαι βέβαιος. Βαντεκάμπ, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ως μέλος ε, της ομάδας του ΕΛΚ και της Επιτροπής Μεταφορών και ως Ολλανδός, καλώς ορίζω το σχέδιο της Επιτροπής Γιούνκερ. Συχνά δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο Eckhout. Στην προκειμένη περίπτωση όμως πρέπει να πω ότι στην Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και όχι μόνο τις απειλές γιατί για πολύ καιρό σκεφτόμασταν μόνο τις απειλές. Τώρα θα πρέπει να δούμε και τις προκλήσεις που κρύβονται. Να σας πω όμως ότι το ιδανικό ε, μονοπάτι αντιμετωπίζει διάφορες εμπόδια. Ένα από τα εμπόδια είναι ότι το Connecting European Facility στον τομέα των μεταφορών δίνει περίπου το μισά από τα χρήματα, από τους πόρους. Αυτό το κάνουμε όμως ε, με κάθε ευχαρίστηση και με τον Ολλανδικό τρόπο, γιατί θεωρούμε ότι θα υπάρξει συντελεστής πολλαπλασιαστικός και για κλασικές υποδομές. Καταλαβαίνω ότι το διαδίκτυο και η Ενεργειακή Ένωση χρειάζονται πολλά χρήματα και πολλούς πόρους, αλλά θέλουμε να προωθήσουμε και τις κλασικές υποδομές. Θα είναι μία πρόκληση προκειμένου να πιστεί ο ιδιωτικό κλάδο για το σχέδιο Juncker. Κοιτάξτε και τα επιτόκια. Και μία ερώτηση να κάνω προ το Συμβούλιο. Πόσα χρήματα έχει ζητήσει ήδη ο πρόεδρο του Συμβουλίου από τα κράτη-μέλη για να υποστηρίξει το σχέδιο Juncker. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα η κυρία Καλοζεμπάλ Ρουμπιέλ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο Κατάνεν. Δεν έχει λειτουργήσει η λιτότητα στην Ευρώπη και γι' αυτό ζητάμε να υπάρξουν βαθιές και σημαντικές αλλαγές. Και γι' αυτό νομίζω ότι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προγίνει προς τη σωστή κατεύθυνση επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ένα ισχυρό, το ισχυρότερο μέσο το οποίο έχει τη διάθεση της Ευρωπαϊκή Ένωση για να μεταρρυθμίσει την οικονομία της. Δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα βέβαια, αλλά και η ποιότητα των προγραμμάτων τα οποία θα υποστηριχθούν. Ζητάμε λοιπόν ένα διαρθρωμένο γύρω από την Ευρώπη και τις πραγματικές της ανάγκες πρόγραμμα επενδύσεων έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη και η αηφορία στην ανάπτυξη. Για μια ακόμη φορά λοιπόν ότι θα λέγουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα στους πολιτικούς στόχους και στα οικονομικά μέσα γιατί δεν θα μπορέσουμε σε καμία περίπτωση να εφαρμόσουμε τη στρατηγική μας με τον σημερινό προϋπολογισμό και με τα σημερινά επενδυτικά προγράμματα. Όπως είπα όμως πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Απαιτείται το πρόγραμμα αυτό να λειτουργήσει και να λειτουργήσει σωστά για να αναζωογονήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα πρέπει να εκπληρώσουμε πάρα πολλά κριτήρια. Καταρχάς το κριτήριο της προσθετικότητας είναι σημαντικό. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να το χρηματοδοτήσουμε αν δεν έχει πραγματική ε, προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Και θα πρέπει επίσης ε, να έχει και συγκεκριμένα αποτελέσματα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Και ε, ιδιαίτερα ξέρετε ότι οι αγορές αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα σε επίπεδο ε, επενδύσεων. Υπάρχουν πάρα πολλά που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προγραμμάτων αυτών έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά. Θα ήθελα εδώ να απευθύνω μια έκκληση προς το Συμβούλιο και όλες τις χώρες να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα αυτό έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί επαρκώς και να υπάρχει το κεφάλαιο που θα βοηθήσει τη βελτίωση των επενδύσεων. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ένα λεπτό και μισό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, πολλά είναι τα ανοιχτά ερωτήματα γύρω από το πακέτο Γιούνκερ και μακάρι να είχαμε και κάποιες απαντήσεις. Το Ευρωκοινοβούλιο να δώσει 8 δισεκατομμύρια και μετά ξεμπερδέψαμε, λέει. Αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι trust fund. Δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοση λογαριασμών. Δεν θα έχουμε επομένω ποτέ λόγο για τους κινδύνους. αλλά θα έχουμε χάσει τα 8 δισεκατομμύρια από τον δομέα της έρευνας. Υπάρχουν ερωτήματα, γιατί αυτοί που έχουν τις εμπειρίες μέχρι τώρα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ως μέλος της ε, Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, μπορώ να σας πω ότι για το 2007 έως 2013 μόνο 40% 40% των κονδυλίων που διαθέσαμε για χρηματοδότηση έργων έφτασαν στον τελικό δικαιούχο. Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο επειδή έχουμε τώρα το πακέτο. Έχω λοιπόν πολλές ερωτήσεις και χρειάζομαι απαντήσεις. Θέλω να πω ακόμη. Αρκεί να δίνουμε λεφτά. Η Ελλάδα έχει την χαμηλότερη απορροφητικότητα των χωρών της Μεσογείου. Υπάρχουν περιφέρειες που δεν μπορούν καν να διαχειριστούν έργα. Άρα χρειάζεται όχι μόνο χρηματοδότηση, αλλά και παροχή τεχνικής βοήθειας. Ε, έγινε και, τέτοιο και ένα ερώτημα. Τι προσφέρουμε στους επενδυτές ο DAX στη Γερμανία ανέβηκε τα τελευταία χρόνια συν 95%. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε επενδύσεις που να τις πληρώσουν ακριβά τελικά οι χρήστες τους. Ευχαριστώ. Κύριε Βανίστελ Ρόι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και υποστηρίζω απόλυτα το σχέδιο Juncker για τις επενδύσεις και για την πραγματική οικονομία. Αλλά παρόλα αυτά έχω να κάνω κάποιες προτερήσεις. Πρώτον, πιστεύω ότι Μιλάμε για 460 δισεκατομμύρια πραγματικά πραγματικές αξίες. Η σχέση που υπάρχει με την απόδοση είναι πολύ ασαφής. Πρέπει να κάνουμε πιο πολλά. Εμείς έχουμε πάρα πολλά τέτοια προγράμματα. Έχουμε εμπειρία. Πολλά μπορούμε να κάνουμε με τα εφιστάμενα χρηματοοικονομικά μέσα στους προπολογισμού μας. Κατά δεύτερον, Χαίρομαι για τη θέματα προστατικότητας και συμπληρωματικότητας. Θα πρέπει να φροντίσουμε το χρέος το οποίο υπάρχει αποκεντρωμένα σε διάφορα έργα να αναλυφθεί από την ΕΤΕΠ και τελικά να μην υπάρξουν επιπλέον επενδύσεις. Μία ερώτηση προς το Συμβούλιο και προς εσάς. Τα κριτήρια είναι πάρα πολύ ασαφή σε τελική ανάλυση. Σε περίπτωση που τα πράγματα εξελιχθούν ως εξή, τα χρήματα τελικά καταλήξουν στα παλαιά κρατημέλη και δεν θα φτάσουν στα νέα κράτη-μέλη. Θα θεωρήσουμε ότι αυτό είναι αποδεκτό. 80, 90% δηλαδή σε κάποια κράτη-μέλη και όχι σε κάποια άλλα. Γι' αυτό μιλάμε. Και να τονίσω και τα, για τα διασυνοριακά έργα, γιατί εκεί χρειάζεται η Ευρώπη ιδιαίτερως και αυτά τα project, αυτά τα έργα θα έχουν προτεραιότητα. Εδώ θα θέλω να απαντήσει το Συμβούλιο, αν γίνεται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρας, για 1,5 λεπτό. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην Ευρώπη έχουμε υψηλή ανεργία, πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, απειρχιωμένες δομές, λίγες επενδύσεις, μικρή ανταγωνιστικότητα και πολύ χαμηλή ανάπτυξη και απασχόληση. Το σχέδιο που υποβάλλεται σήμερα αποτελεί μια μόνο πρωτοβουλία και μάλιστα συμπληρωματικού χαρακτήρα το νέο σας σχέδιο ακολουθεί νέο δρόμο, νέος δρόμος. Αυτό με ικανοποιεί. Αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο για όλα τα εφιστάμενα μέτρα τα οποία είχαμε ήδη εγκρίνει. Πρέπει να είναι μια πρόσθετη πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Χρειάζεται μια πρωτοβουλία για μια ευρωπαϊκή επενδυτική επίθεση. Η ιδέα που θα κρύβεται από πίσω και χρειαζόμαστε έργα τα οποία να είναι βιώσιμα επιτυχή. Γιατί αλλιώ δεν πρόκειται να προσελκύσουμε ιδιώτε επένδυτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι συνυπεύθυνο. Αυτό θα το δείξουμε μέσα από τις εκθέσεις μας και την εργασία μας και στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά ιδίως στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ε, γι' αυτό όμως χρειαζόμαστε τον διάλογο. Δεν μας αρκεί να είμαστε οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση των επενδύσεων. Οι χώρες μέλη θα πρέπει να διπλασιάσουν το Ταμείο και με χρήματα και με εγγύσεις. Διακόπτει τώρα η κυρία Πρόεδρος. Ο κύριος Έλερ, ένα λεπτό και 30 δεύτερα. Κύριε Κατάινεν, Είπε ο Μάνφρετ Βέιμπερ θα σας υποστηρίξουμε. Είναι σωστό το project αυτό. Χρειάζεται και η σωστή δόμηση. Ερωτήσεις. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του ΕΦΣΥ σε σχέση με τα εφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα Horizon 2020 κλπ. Έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και πώς μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία αντί να ανακατευθύνουν της ε, τις Δεύτερο, τι είδους προφίλ κινδύνου αναζητούμε. Να το πω διαφορετικά. Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο μόχλευσης. Αυτό είναι σημαντικό. Διότι υπάρχουν ήδη χρηματοδοτικά εργαλεία. Και τέλος, αντί να πάρουμε τα χρήματα από την έρευνα και την, και την ε, ανάπτυξη, είναι καλύτερα να τα πάρουμε από αλλού. Merci. Σας ευχαριστώ. Θα προχωρήσουμε τώρα στο τμήμα της συζητήσεως Catch the Eye. Η κυρία Μάλετιτς, ένα λεπτό παρακαλώ. Ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Αντιπρόεδρο και θα ήθελα να πω ότι ένα σημαντικό μάθημα της επενδυτικής πολιτικής από την πολιτική συνοχής που αποτελεί και ένα μέσο ανάπτυξης και επενδύσεων. Ένα σημαντικό λοιπόν μάθημα είναι ότι θα πρέπει όλες οι δυνάμεις μας να υποστηρίξουν τα ποιοτικά προγράμματα και την ενίσχυση των ανθρωπινών πόρων. Αυτά λείπουν στα ευρωπαϊκά έργα και οι ανθρώπινοι πόροι όμως. Εδώ θα έπρεπε να εστιαστεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποιούν τα ταμεία συνοχής θα έπρεπε να επενδύσουν σημαντικά και στην συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών. Ελπίζω η νέα επενδυτική πολιτική να μην αντικαταστήσει την ε, πολιτική συνοχής, αλλά να αποτελέσει συμπληρωματικό παράγοντα, προκειμένου οι χώρες αυτές να έχουν ε, την δημοσιονομική ενίσχυση και να μην χρειαστεί να σταματήσουν επενδύσει, αλλά να αξιοποιήσουν στο πλήρες το δυναμικό του. Ευχαριστώ, κυρία Γέλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Εμεί ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιούμε για τι μεταφορέ ε, το μέσο Connecting Europe, το οποίο βελτιώνει τι ε, υποδομέ και δημιουργεί θέσει απασχόληση. Ε, το θέμα είναι ε, ότι θα το εγκαταλείψετε αυτό για να περάσετε στο πρόγραμμα επενδύσεων του Juncker ε, και θα τα χρησιμοποιήσετε για προγράμματα μεταφορών και με τον Ευρωπαϊκό Έλεγχο βέβαια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου ελπίζω. Γιατί ξέρετε τι έγινε με το πρόγραμμα Κάστορ που ήταν ένα από τα πρότυπα προγράμματα και το οποίο όπως γνωρίζετε δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και θα πρέπει παρόλα αυτά να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά με σωστό έλεγχο από πλευρά των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Η ε, κυρία Φόρτ, συνάδελφοι, χρειαζόμαστε επενδύσεις, χρειαζόμαστε επενδύσεις του ιδιωτικού κλάδου και οι επιχειρήσεις, οι μικροεπιχειρήσεις θα πρέπει να ξέρουν ότι είμαστε στο πλευρό τους. Έχω γεμίσει στο, από ηλεκτρονικά μηνύματα από επιχειρήσεις που έχουν σταματήσει το εμπόριο τους στον πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας μας, της ψηφιακής επιχειρηματικότητα. Αυτά τα προγράμματα θα είναι για τις μεγάλες επιχειρήσεις που προσπαθούν να αποφεύγουν τους ε, φόρους, αλλά είναι υπερβολικά δαπανηρά για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν απαραίτητα στην ε, ψηφιακή εποχή. Συμβούλιο, σε εσά είναι το μπαλάκι. Μην ε, περιοριστείτε μόνο στις σκέψεις και σε λόγια, γιατί δεν θα σας πάρουν στα σοβαρά συμβούλιο. Σας παρακαλώ, δώστε ε, απαλλαγή στις μικρές επιχειρήσεις. Απλά κάντε το. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Γιάκοφτσίτς για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Ε, η ιδέα αυτή θα κρίνει την ιστεροφημία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εντολή που δίδουμε εμείς στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, θα χαρακτηριστεί επίσης από τις δυνατότητες επιτυχίας και αποτυχίας και γι' αυτό θα ήθελα εκ των προτέρων να πω ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση Δέχομαι βέβαια και αναγνωρίζω τις κριτικές και θα πρέπει να τις συζητήσουμε, αλλά ας προτείνουμε εναλλακτικέ λύσεις. Πού είναι αυτές οι λύσεις, δεν ακούγεται τίποτα. Συνεπώς πιστεύω ότι μια ολόκληρη σειρά προγραμμάτων θα πρέπει να επιλεγούν σε συνέργεια με τα κράτη-μέλη, με τις περιφέρειες, με τα ιδιωτικά κεφάλαια, γιατί μόνον τότε και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ελπίζουμε μια κάποια επιτυχία. Βιέγας, ένα λεπτό. Ευχαριστώ αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις. Καλύπτει μια κρίσιμη ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, την έλλειψη ανάπτυξης, και απαιτούνται βέβαια μορφές χρηματοδότησης για να μπορέσει να λειτουργήσει το ταμείο αυτό και γι' αυτό ε, προσπαθούμε να προσελκύσουμε υπεύθυνου επενδυτές. Είναι μια ανάγκη που θα συνεχίσουμε να την νιώθουμε και στο μέλλον, βασίζεται στη συνεργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Οι ιδιώτες θέλουν να υπάρξουν κέρδη, το δημόσιο θέλει να αποσβέσει τις επενδύσεις του δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επενδυτές, αλλά δεν υπάρχουν επενδυτές που να έχουν εμπιστοσύνη στο παρόν κλίμα. Απαιτείται να υπάρξει λοιπόν ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που να καλύψει τις ανάγκες της συνοχής στο κοινωνικό επίπεδο. Βάλει ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ όπως υπόθηκε και από τους συναδέλφους εκφράζω τις ανησυχίες μου γιατί τα κεφάλαια αυτά, οι πιστώσεις αυτές φεύγουν από προγράμματα της έρευνας και θα περάσουν σε προγράμματα για τις υποδομές όπου θα καλύψουμε εκεί τις ανάγκες οργανωμένων συμφερόντων και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ξέρετε τι έγινε πρόσφατα στο Λουξεμβούργο και ίσως γι' αυτό να υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα Juncker να δοθεί ένα άλοθη στους σοσιαλιστές οι οποίοι εγκαταλείπουν την μάχη εναντίον της λιτότητας ε, και έχουν κοροϊδέψει τους εκλογείς τους από τις πολιτικές που τις υπεσχέθηκαν κάποια σοσιαλιστικά κόμματα δήθεν για να καταπολεμήσουν τη λιτότητα. Λοιπόν είναι επικίνδυνο το πρόγραμμα αυτό και ακριβώς ε, διατρέχουμε τον κίνδυνο να διαψεύσουμε τις προσδοκίες του πολίτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχέδιο Juncker παρουσιάζεται από πολλούς ε, σαν το θαυματουργό όπλο. 315 δισεκατομμύρια ευρώ. Να δούμε όμως τι θα γίνει 21 ε, δισεκατομμύρια προέρχονται από την ευρωπαϊκό προπολογισμό και περιμένετε 15 του συντελεστή. Δεν είναι, ξέρετε όμως, θαυματουργό αυτό το όπλο, αυτό το μέσο. Μάλλον ε, ε, περιμένουμε θαύματα από ένα τέτοιο μέσο. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη ευθύνη. Θα έπρεπε το κράτος να, έχει, να δίνει την εγγύηση στην Ουγγαρία έχουμε πάρα πολλέ αρνητικέ εντυπωσει και εμπειρίε από τη συμπράξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Γιατί τελικά ποιο είναι ο στόχο οι θέση απασχόληση. Οι θέση απασχόληση όμω σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από τι μικρομεσαίες επιχειρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό αυτού πρέπει να υποστηρίξουμε κάθε επιγόντος. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόγκοβιτς για ένα λεπτό. Oh, Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το Ταμείο Επενδύσεων πρέπει να είναι χρήσιμο ιδιαίτερα. Ε, επίσης να στηρίξουμε και τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας γιατί αυτά θα οδηγήσουν σε περισσότερες θέσεις απασχόλησης και σε μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ζητώ από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο να συνεργαστούν με τις χώρες μέλη για να αποφύγουμε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Να διαπιστώσουμε δηλαδή ότι στο τέλος του προγράμματος ότι τα προγράμματα αυτά επιστρέφουν στις πλούσιες χώρες. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές καθυστερήσεις ακριβώς λόγω της έλλειψης των ιδιωτικών κεφαλαίων. Ας είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε το ταχύτερο δυνατόν τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, όχι μόνο σε επίπεδο ένωσης, αλλά και στα κράτη-μέλη. Πρόεδρε, το πακέτο που προτείνει ο Επίτροπος Κατάνιν είναι σημαντικό βήμα, αλλά η δική μου ομάδα το ζητάει αυτό εδώ και χρόνια και λέει ότι χρειαζόμαστε πιο πολλέ επενδύσει, γιατί μόνο τα μέτρα λιτότητα είναι σαφέ ότι από μόνα του δεν φτάνουν για την ανάπτυξη. Καλωσορίζω λοιπόν την νομοθετική αυτή πρόταση σε ό,τι αφορά το ταμείο αυτό, αλλά πιστεύω ότι από εμά εξαρτάται να λειτουργήσει. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή εφαρμογή. Από εμά εξαρτάται. Για να το πετύχουμε όμω αυτό, θα πρέπει πολλά να κάνουμε και να δουλέψουμε σκληρά. Τα βασικά στοιχεία, πέρα από αυτά που έθεσαν οι συνάδελφοι, για την επιλογή των σωστών έργων, είναι κρίσιμα στοιχεία αυτά. Να υπάρχει προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, να μην είναι έργα τα οποία έτσι και αλλιώ θα ε, είχαν χρήματα. Και ίσως λοιπόν τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να δίνουν τα χρήματα αυτά με βέλτιο τρόπο στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω όμως είναι ποιος θα αποφασίσει για τα έργα αυτά. Είπατε ότι το Κοινοβούλιο θα έχει ένα ρόλο στις ακροάσεις. Θα έχει νόημα όμως ε, η συμμετοχή του Κοινοβουλίου για την επιλογή. Σας ευχαριστώ. Εδώ λίγη το Catch the Eye. Δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Κατάινεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την συζήτηση, ευχαριστώ για τις ιδέες που υποβάλατε. Θέλω να τονίσω την, τον βασικό χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου το επενδυτικό σχέδιο δεν θα αλλάξει τα πάντα μόνο του. Χρειαζόμαστε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, χρειαζόμαστε δημοσιονομική πολιτική που να αποκαθιστά την εμπιστοσύνη, χρειαζόμαστε πολιτικές παρακολούθησης, monitoring δηλαδή, και χρειαζόμαστε και πανευρωπαϊκές δράσεις για να ενθαρρύνουμε ιδίω τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στην Ευρώπη. Για αυτούς τους λόγους το σχέδιο επενδύσεων δεν είναι ένα εφάπαξ μέτρο παροχής κινήτρων, είναι μια διαρθρωτική ευρωπαϊκή απάντηση με τρεις πτυχές. Πρώτον, έχει ένα ταμείο ανάληψης κινδύνου, ένα risk fund, για να ενθαρρύνει τους επενδυτές να πάνε να επενδύσουν σε χώρες με μεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο, περιφέρειες κλπ. και ιδίως σε μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Δεύτερη πτυχή είναι ο διαφανής αγωγός, transparent pipeline δηλαδή, που θέλουμε σε αυτόν να προωθήσουμε έργα ώστε το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο να μπορεί να επιλέξει. Αυτό το ζητούν και οι θεσμικοί επενδυτές και οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα. Λένε ότι η καθημερινή μας δουλειά είναι να επενδύουμε στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκουμε αρκετά βιώσιμα και καλά διαρθρωμένα επενδυτικά έργα που να μπορούμε δηλαδή να πάμε να επενδύσουμε σε αυτά. Θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε και τον ιδιωτικό τομέα αλλά και το δημόσιο τομέα να διαρθρώσουν τα σχέδια αυτά, τα project αυτά. Ενισχύουμε λοιπόν την τεχνική συνεργασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ώστε όλα τα τμήματα της Ευρώπης να υποφεληθούν από τις πρωτοβουλίες αυτές. Και η τρίτη πτυχή που κατά τη γνώμη μου είναι και η πιο σημαντική του σχεδίου επενδύσεων είναι η πτυχή της ενίας αγοράς, διότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή διαρθρωτική μεταρρύθμιση που μπορεί να δημιουργήσει νέες αγορές, νέες ευκαιρίες και για μικρές μεσαίες αλλά και για μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Και εκεί the sky is the limit για την δημιουργία θέσεων, νέων θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό πρέπει νομίζω όλοι να στοχεύσουμε στην πτυχή αυτή της ενιαίας αγοράς χωρίς να μην τη λησμονούμε. Παρόλο βέβαια που τα χρήματα, τα κονδύλια έχουν μεγάλη ελκυστικότητα, αλλά η ενιαία αγορά είναι αυτή που μπορεί να ωφελήσει περισσότερο. Όσοι εξ ενδιαφερόμαστε να ενισχύσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ενδιαφερόμαστε να δώσουμε περισσότερα από δημόσιους πόρους σε χρηματοδότηση μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Αυτούς λοιπόν σας ενθαρρύνω να δείτε τι κάνει η Ισπανική κυβέρνηση και ενθαρρύνω και κάθε χώρα να το κάνει. Χρησιμοποιούν τα κονδύλια των διαρθωτικών ταμείων ως χρηματοδοτικό εργαλείο, προσφέρουν λοιπόν έτσι περισσότερη ρευστότητα στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος χρήσης των διαρθωτικών ταμείων. Αν θέλετε να δώσετε περισσότερα δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία που μένει ακόμα άθιχτη σε πολλές χώρες μέλη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περάσει το μήνυμα αυτό σε όλες τις χώρες μέλη. Ας μην λησμονούμε ότι η αρχική ΕΤΕ θα συνεχίσει να ε, λειτουργεί, θα δίνει 60 με 70 δισεκατομμύρια το χρόνο σερεστότητα και χωρίς τις συνεισφορές των χωρών μελών. Ο λόγος για τον οποίο το νέο ταμείο είναι μικρότερο είναι διότι στοχεύει σε έργα υψηλού κινδύνου. Δεν γνωρίζουμε τι είδους ζήτηση, πόσο μεγάλη ζήτηση υπάρχει για τέτοιου είδους κονδύλια. Όμως κυρίες και κύριοι αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω πράγματι να συνεργαστούμε πολύ στενά όταν θα πάρουμε χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε το ίδιο ε, ποσό χρημάτων, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Άρα και η έρευνα θα λάβει περισσότερα χρήματα όταν χρησιμοποιήσουμε το εφέ της μόχλευσης. Θα μπορούμε λοιπόν να κινηθούμε ταχύτατα μαζί για να εκμεταλλευτούμε και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας, για τους πολίτες. Χρειαζόμαστε δουλειές. Αυτό είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο θεσπίζουμε το νέο αυτό επενδυτικό σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος κύριος Βίλαντ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Θα λάβει το λόγο η Υφυπουργός κυρία Καλνίνια Λουκασέβιτσα. Αξιότιμα μέλη, Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη συζήτηση που προηγήθηκε και η οποία απέδειξε τη σημασία την οποία δίδουμε σε αυτού του νέου τύπου επενδύσεις στην Ευρώπη μετά από χρόνια στασιμότητας. Αποδεικνύεται η αποφασιστικότητα των θεσμικών οργάνων να ολοκληρώσουν ένα πετυχημένο επενδυτικό πρόγραμμα που θα επιτρέψει την αηφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής έλαβα υπόψη μου πέντε ε, τομείς ερωτήσεων που τέθηκαν. Πρώτον, το θέμα της γραφειοκρατίας και της ανάγκης για τη μείωση αυτής. Μετά τέθηκε το θέμα των πηγών επενδύσεων και για τη διασύνδεση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τρίτον, και έχει μεγάλη σημασία, υπογραμμίστηκε η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι επενδύσεις αυτές δεν θα πρέπει να ωφελούν μόνο τους επενδυτές αλλά τους πολίτες και τους εργαζομένους και τέθηκαν επίσης και ερωτήσεις ε, η λεγόμενη χρήση ευφυών μορφών επενδύσεων και αηφόρων επενδύσεων και τέλος επίσης ε, θέματα δημοκρατικού ελέγχου ευθύνη και συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαχείριση του Ταμείου αυτού. Θα ήθελα να αναγνωρίσω φυσικά τώρα την σημασία αυτών που είπε ο κύριος Βέμπερ, ο κύριος Καμάλ και η κυρία Ροντρίγες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρίτο πυλώνα του επενδυτικού αυτού στρατηγικού προγράμματος. Όπως είπα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, ίσως ο τρίτος πυλώνας είναι αυτός ο οποίος τελικά θα παίξει τον σημαντικότερο ρόλο για την ενίσχυση των ε, επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή των τριών πυλώνων είναι μια σωστή επιλογή που θα ανεβάσει το επίπεδο των επενδύσεων. Είναι κάτι το πολύ θετικό και μακροπρόθεσμα, αλλά είναι αρκετά περίπλοκο σαν θέμα σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Και γι' αυτό όχι μόνο θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε το ταμείο αυτό, αλλά να απομακρύνουμε και τα εμπόδια εκμεταλλευόμενοι την εσωτερική αγορά, ιδιαίτερα στον τομέα της Ένωσης της Αγοράς Ενέργειας, της ε, ψηφιακής οικονομίας κτλ. Πολλά μπορεί να γίνουν λοιπόν και σε εθνικό επίπεδο. Τώρα για τις πιθανές επενδύσεις ε, συμμετοχές των κρατών μελών ε, στο Ταμείο. Ε, δεν έχουμε ακόμα καταλήξει στις ε, τελικές λεπτομέρειες. Τώρα έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε την ομοθετική πρόταση, αλλά στόχος μας είναι ότι οι νέες αυτές επενδύσεις ε, μπορεί να δημιουργηθούν. Είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη και οι εθνικές επενδυτικές τράπεζες θα πρέπει να μπορούν να συνεισφέρουν στο Ταμείο. Αυτό είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούν τα κράτη-μέλη να επενδύσουν αυτού του τύπου τις επενδύσεις. Μπορούν να παρεμβαίνουν και σε επίπεδο προγράμματος ή στις ευρύτερες πλατφόρμες, τις επενδυτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπολογίζουν ότι το επίπεδο επενδύσεων το οποίο υπολογίζεται να κινητοποιηθεί θα φτάσει τα 315 δις νέων ε, πιστώσεων. Πολλά από αυτά θα έρθουν από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ε, έχει στη διάθεσή του μια κάποια ρευστότητα, είναι πραγματικά χρήματα και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό βέβαια θα συμπληρωθεί και από ε, συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις από τα κράτη-μέλη και αυτό θα αυξήσει το τελικό ποσό. Όταν μιλάμε για την προστιθέμενη αξία του Ταμείου, να υπογραμμίσω ότι στόχος είναι η διευκόλυνση νέων μορφών επενδύσεων. Το θέμα είναι να μην αποκλείσουμε αλλά να προσελκύσουμε τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα πάντως έχουμε εξετάσει τις λεπτομέρειες της πρότασης και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σύντομα. Βασικό χαρακτηριστικό της πρότασης αυτής είναι η απροσθετικότητα. Θα πρέπει να στηρίξουμε προγράμματα τα οποία είναι εκτός χρηματοδοτήσεων. Προγράμματα τα οποία θεωρούνται πολύ επικίνδυνα σε επίπεδο επενδυτικών κεφαλαίων. Πρέπει λοιπόν να ε, δώσουμε τις απαιτούμενες εγγυήσεις και να προσελκύσουμε τους ιδιώτες. Ο κύριος Μπούλμα έθεσε πολύ σημαντικά θέματα στα οποία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες απαντήσεις κατά τη διάρκεια των εσωτερικών και των διαθεσμικών συζητήσεων. Τα χρήματα θα πρέπει να πάνε εκεί όπου πραγματικά χρειάζονται και θα πρέπει να έχουν σαν στόχο τη διασφάλιση υψηλότερου επίπεδου βεβαιότητας για τους επενδυτές. Φυσικά, το Ταμείο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα θέματα της ανισότητας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Αυτός είναι ο βασικός του στόχος. Και έτσι θα μπορέσουμε βραχυπρόθεσμα να στηρίξουμε τη ζήτηση και να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης της Ευρώπης ε, μέσω μακροπρόθεσμα. Η απασχόληση είναι στόχος πάντως κομβικός. Η αύξηση των επενδυτικών δυνατοτήτων θα βοηθήσει λοιπόν την αγορά εργασίας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπουμε λοιπόν να στηρίξουμε και τις μεθόδους χρηματοδότησης των μικρομεσαίων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, διότι συνεισφέρουν τα μάλλα στην καταπολέμηση της ανεργίας στην Ευρώπη. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοήσουμε, γιατί χρειαζόμαστε να στηρίξουμε τη δραστηριότητα των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων. Σχετικά τώρα με το περιεχόμενο των συζητήσεων στο Συμβούλιο, να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι η χθεσινή συζήτηση στο ΕΚΟΦΗΝ έγινε δημόσια Νομίζω ότι κάποια στοιχεία θα σας ε, δείξουν ποιο ήταν το περιεχόμενο. Οι Υπουργοί ε, είπαν ότι είναι αποφασισμένοι να καταστήσουν το πρόγραμμα αυτό επιτυχές. Συμφωνούν ότι πρέπει να βοηθηθούν αυτά τα προγράμματα τα οποία απαιτούν περισσότερες εγγυήσεις. Τα προγράμματα τα οποία δημιουργούν όμως θέσεις απασχόλησης και μεταφέρουν την τεχνολογία στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στις περιοχές που παρουσιάζουν μια κάποια υστέρηση. Τέθηκε και το θέμα της προσθετικότητας σαν βασικό κριτήριο. Υπάρχουν πολλά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε τα θέματα αυτά να τύχουν λύσεων. Οι συζητήσεις που θα ακολουθήσουν δεν θα είναι εύκολες στο Συμβούλιο, πάντως νομίζω ότι θα δώσουν καλά αποτελέσματα. Τώρα για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόταση δημιουργίας του Ταμείου, έτσι ώστε να συμφωνήσουμε το ταχύτερο δυνατόν και να επιτρέψουμε τη ροή ε, ρευστότητα στις οικονομίες μας. Απαιτείται βέβαια να σεβαστούμε ορισμένες βασικές αρχές όπως ε, η δημοσιοποίηση ε, και ο έλεγχος ε, της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η ελεύθερη αδέσμευτη επιλογή προγραμμάτων. Το Συμβούλιο θα πρέπει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να εξετάσει τις προτάσεις αυτές. Νομίζω ότι μπορούμε να σεβαστούμε τις προθεσμίες τις οποίες έχει ορίσει το Συμβούλιο χωρίς έτσι να μειώσουμε ή να υπονομεύσουμε την ποιότητα της νομοθετικής ρύθμισης. Νομίζω ότι μπορούμε με τον τρόπο αυτό να πετύχουμε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο. Οι πολίτες περιμένουν να αναλάβουμε δράση τάχιστα, δεν έχουμε χρόνο. Αγαπητά μέλη λοιπόν να συνεργαστούμε έτσι ώστε πράγματι το επενδυτικό αυτό ταμείο να τεθεί σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν. Ας αφήσουμε πίσω μας την οικονομική κρίση, ας αφήσουμε πίσω μας τις προσπάθειες, την αδράνεια μάλλον του παρελθόντος. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ παρά κυρία Καλινάζου Λουκασεβίκα. Και έτσι ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση.